morning, dear colleagues. Thank you for being here. Thank you for your patience. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Είχαμε τη συνεδρία των συντονιστών στις 9, βγήκε σε μία ώρα, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην ε, τακτική συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σας καλωσορίζω όλους ε, και θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε χτες στο σημείο 8 που είναι η μελέτη σχετικά με τις πολιτικές των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα παιδιά με αναπηρία. Εδώ θα ακούσουμε την παρουσίαση της κυρίας Μάρτα Μπαγιαστέρος και της κυρίας Ναταλή Μεράς από του Μιλιές της Βρυξέλλες. θα παρουσιαστεί μελέτη σχετικά με τις πολιτικές ε, των κρατών μελών για τα παιδιά με ανεπηρίες που ζήτησε η ΛΥΜΠΕ από το Τμήμα Πολιτικής για να αξιολογηθεί η κατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών με ανεπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη για νομοθεσία και λήψη μέτρων. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μέρενς για τις παρουσιάσεις ε, και κατόπιν ε, θα προβούμε σε συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Μέρενς. Καλημέρα σας. Λέγομαι Νατελμερένης από τη Μιλιέ που ε, είναι ένα γραφείο περιοχής βουλών για θέματα ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα παρουσιάσω εδώ θέματα που αφορούν την πολιτική των κρατών μελών ε, για παιδιά με ανεπηρίες. Η μελέτη έχει στόχο να αξιολογήσει την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την κατάσταση. Έτσι λοιπόν από την αρχή θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μία ρητή αρμοδιότητα για το θέμα των παιδιών με εμπειρία, αλλά έχει το ρόλο να προωθήσει τα δικαιώματα των παιδιών και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις Η μελέτη εξέτασε 18 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Μάλτα μέχρι τη Φιλανδία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, το Ενωμένο Βασίλειο και ήθελε να καλύψει ευρέως ε, το ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι κάναμε για τη μελέτη. Εξετάσαμε τη σύμβαση του ΙΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και για τα άτομα με ανεπηρίες και εκεί εντοπίσαμε ποια είναι τα δικά δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίε. Κατόπιν εξετάσαμε την νομοθεσία των 18 κρατών μελών και θέλαμε να εξετάσουμε αν εγγυούνταν τα δικαιώματα αυτά όπως μπορείτε να δείτε, τα δικαιώματα είναι τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, δικαίωμα ε, σε ακρόαση, δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, δικαίωμα σε ένταξη κτλ. Επίσης είδαμε και τις πρακτικές εφαρμογής. Ε, τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας έδειξαν ότι σε όλα τα 18 κράτη-μέλη υπήρχε σχετική νομοθεσία για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών ανεπηρίας, όμως υπήρχε πρόβλημα στην πρακτική εφαρμογή. Επίσης, ε, είδαμε σαφές ότι η οικονομική κρίση έχει αντίκτυπο στην κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες σε ό,τι αφορά το κόστος του προϋπολογισμού για την παροχή υποστήριξη στα παιδιά και στην οικογένεια. Τώρα, θα σας παρουσιάσω δύο παραδείγματα σήμερα για να δείτε πώς είναι η κατάσταση για τα παιδιά με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο παράδειγμα έχει να κάνει με το δικαίωμα σε μη εισαγωγή διακρίσεων βάσει της αναπηρίας. Ενώ σε όλα τα κράτη-μέλη υπήρχε εγγύηση δικαιωμάτων για να μην υπάρχουν διακρίσεις βάσει της αναπηρίας σε πολλά κράτη-μέλη αυτά τα δικαιώματα αφορούσαν μόνο τομείς όπως είναι οι μεταφορές, η παιδεία, η υγεία και ε, ξέρετε ότι σε κάποιους τομείς ε, δεν ήταν σχετική αυτή η τομή για τα παιδιά. Πιο σχετική είναι η εκπαίδευση, η πρόσβαση στην υγεία κτλ. Βλέπουμε επίσης ε, ότι ε, μια ε, απαραίτητη στέγαση η στέγαση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών και επίσης πρέπει τα παιδιά να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα παιδιά. Για να γίνει αυτό χρειάζεται κάποια προσαρμογή. Δηλαδή, αν ένα παιδί είναι σε καροτσάκι, θα πρέπει όλα τα μαθήματα να γίνονται στο ισόγειο παραδείγματο χάρη του σχολείου. Επίσης είδαμε ότι δεν ήταν κατανοητή αυτή η έννοια από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή από το γενικό κοινό. Παραδείγματο χάρη ένα παιδί με δυσλεξία έχει δυσκολία να διαβάσει και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για τις εξετάσεις όταν ε, οι γονείς ζητούν περισσότερο χρόνο για τις εξετάσεις, ένα άλλο παιδί, άλλες οικογένειες ε, θεωρούν ότι αυτό είναι προνόμιο παρά μια διευκόλυνση. Επίσης, η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντική για το παιδί, η προσβασιμότητα σε κτίρια, σε δημόσιες μεταφορές και σαφώς έλειπε σε πολλά κράτη-μέλη. Ως αποτέλεσμα, προτείναμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε η έννοια της ε, στέγασης να διευκρινιστεί και να αναλυφθεί δημόσια δράση για να μπορεί να λάβει χώρα μια συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση για την οδηγία κατά της εγωγής διακρίσεων, θέλουμε και ένα εκτιμώντας που να δηλώνει ότι η οδηγία λαμβάνει υπόψη τα παιδιά τις ανάγκες των παιδιών ε, με αναπηρία. Ε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το δικαίωμα σε, στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Δηλαδή τα παιδιά να μπορούν ε, να παρακολουθούν τα μαθήματα στο σχολείο. Όμως σε πολλά κράτη-μέλη δεν αναγνωριζόταν το δικαίωμα σε μια εκπαίδευση ένταξης. Δηλαδή ε, υπήρχε σε πολλά κράτη μέλη αυτή η διάταξη, αλλά δεν υπήρχαν, ε, υπήρχε λήψη πόρη σε ειδικά δημόσια σχολεία. Ένας από τους λόγους ήταν ότι τα σχολεία δεν έχουν το υλικό και τους ανθρώπινους πόρους για να μπορούν να καλωσορίσουν αυτά τα παιδιά. Έτσι λοιπόν το παιδί είτε έχει την επιλογή να πάει σε ένα ειδικό σχολείο ή αν θέλει να πάει σε ένα ε, κανονικό σχολείο. Ε, βλέπουμε εκεί πολλές περιπτώσεις παιδιών που πρέπει να περάσουν τρεις ώρες στο δρόμο μέχρι να φτάσουν σε ένα σχολείο που να είναι κατάλληλο για αυτά. Επίσης, το, προ... το σχολικό πρόγραμμα δεν είναι αρκετά ευέλικτο για να μπορούν να συμμετέχουν στην τάξη παιδιά με αναπηρίε. Και αυτό σημαίνει ότι όταν ε, ένα παιδί πηγαίνει σε ένα μη ειδικό σχολείο, ε, συχνά κάποια παιδιά που έχουν ε, πρόβλημα συμπεριφοράς ή αναπηρίες πρέπει να εγκαταλείψουν το σχολείο γιατί δεν είναι προσαρμοσμένο σε αυτό το πρόγραμμα των μαθημάτων. Επομένως, τι συστήνουμε την ε, ανοιχτή μέθοδο συντονισμού προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές, επίσης να εκπαιδεύσει τους ε, δασκάλους για να καταλάβουν ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και να προωθήσει την ένταξη. Ως γενική σύσταση, θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παροτρύνει τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση για Ανθρώπους με Ανεπηρίες να το πράξουν, καθώς και τα πρωτόκολλα του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Επίσης, θέλουμε το Κοινοβούλιο να προωθήσει την χρήση των πόρων με έναν τρόπο που να προωθούν την ένταξη των παιδιών με αναπηρία στο σχολείο και στην κοινωνία, καθώς και την προσβασιμότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμη για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος, για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να αποτείνουμε τώρα στα μέλη. Υπάρχουν σχόλια, ερωτήσεις. Ο κύριος Αντζελίλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που προφανώς πρέπει να αναλύσουμε επί του συγκεκριμένου. Τρία σημεία θέλω να αναφέρω και είναι τα εξή. Στην πραγματικότητα τα δεδομένα είναι ακόμα ανεπαρκή και μη ακριβή. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι ότι έχουμε περίπου 15 εκατομμύρια παιδιά τα οποία έχουν ειδικέ ε, εκπαιδευτικές ανάγκες. Όμως, από όσο έχω καταλάβει, δεν υπάρχει ακόμα μια στατιστική φωτογραφία ξεκάθαρη, μια στατιστική ξεκάθαρη εικόνα σε ό,τι αφορά τις αναγκαιότητες των παιδιών με ανεπηρίες. Εμείς γνωρίζουμε ότι ένα στοιχείο διάκρισης δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, αλλά και στον αθλητισμό βλέπουμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα και η παροχή ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κάποιες περιπτώσεις, η στήριξη στην οικογένεια, η κοινωνική αρρωγή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, αν υπάρχουν δεδομένα κατά προσέγγιση, γιατί δεν είναι απλό να μελετήσουμε νέες προτάσεις ε, και να απευθυνθούμε στα κράτη-μέλη και να τους ζητήσουμε να υπάρχει και μια στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να ξέρουμε με ακρίβεια ποιες είναι οι προτεραιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω γιατί αυτή η μελέτη είναι εξαίρετο σημείο αφετηρίας. Ευχαριστώ κύριο Στόρβαλτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην πολιτική μου ζωή είμαι ο πρόεδρος μιας ένωσης ε, για ε, ανάπηρα άτομα τα οποία έχουν σωματική ή και πνευματική αναπηρία. Όταν μιλούμε για αξίες ε, στην ομιλία ο πρόεδρος της ε, Κομισιόν ανέφερε το θέμα αυτό και την, το σεβασμό των κοινών ε, αξιών. Όταν λοιπόν αναφερόμεθα στις θεμελιώδεις αξίες, καταλήγουμε σε σλιβερά συμπεράσματα όπως ακούσαμε σήμερα και στο γεγονός ότι δεν έχουμε την συγκεκριμένη αρμοδιότητα να δράσουμε. Έχουμε βεβαίως τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη σύμβαση του ΟΗΕ και ο τρόπος με τον οποίο έχει επικυρωθεί η σύμβαση του ΟΗΕ δείχνει ότι είναι προβληματική. Δεδομένου ότι στα περισσότερα κράτη επικυρώνεται η σύμβαση χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη την ουσία ούτε έχουν την πρόθεση να αλλάξουν την νομοθεσία τους έτσι ώστε να συνάδει με το χάρτη, δηλαδή δεν λαμβάνουν υπόψη το νόημα και δεν εφαρμόζουν την ουσία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει πράγματι να κάνουμε κάτι σοβαρό για να μπορέσουμε να αποκριθούμε στα πρότυπα αυτά, στις ε, ε, υψηλές ε, αξίες τις οποίες όλοι ασπαζόμεσα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Τόβας, η κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και για αυτήν την παρουσίαση. Έχω μια ερώτηση, μάλλον περισσότερο ένα σχόλιο. Αναφερθήκατε σε αυτή την έννοια τη νομική του reasonable accommodation, της ε, εύλογης, του εύλογου δικαιώματος στη στέγαση και νομίζω ότι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι ποιο είναι το καλύτερο περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον, γενικότερα περιβάλλον για ένα, ένα παιδί με αναπηρία. Τόσο για το σχολείο όσο και για τα παιδιά με αναπηρία που θα φοιτήσουν σε αυτό. Γιατί εξάλλου η υψηλή ποιότητα παιδεία είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να ε, έχουν πρόσβαση αργότερα στην αγορά εργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η ανεργία των ατόμων με αναπηρία είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ευρώπη, ακόμα υψηλότερη από τους γενικούς ε, αριθμούς. Πώς, πώς λοιπόν μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτή την υψηλή ποιότητα παιδεία έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και την ένταξη στην αγορά εργασία αργότερα. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από ό,τι φαίνεται. Παρακαλώ. θα επανέλθουμε στην κυρία Μωρέν. Θέλετε να απαντήσετε στα σχόλια ως εδώ. Μάλιστα για να ε, απαντήσω στο πρώτο σχόλιο της κυρίας Αντζελίνη. Είναι σωστό ότι έχουμε έλλειψη στοιχείων, δεδομένων. Στην προσπαθήσαμε για τη μελέτη μας ε, να χρησιμοποιήσουμε και να βρούμε ε, όλων των ειδών τα στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν αλλά πολλές φορές δεν υπήρχαν, διότι πο, πο, για πολλά από τα παιδιά αυτά δεν υπήρχαν στοιχεία ή τα στοιχεία αναφερόντουσαν μόνο στην ηλικία και στο είδος της αναπηρίας. Ε, πράγματι η έλλειψη δεδομένων, ε, η έλλειψη τεκμηρίωσης και στοιχείων είναι ένα πρόβλημα συνεχές και θα θέλαμε να, να έχουμε πολύ περισσότερα. Ε, κυρία Μπαλεστέρος, για να τονίσουμε το θέμα των δεδομένων ε, πολλές φορές δεν υπάρχουν για παιδιά με αναπηρίες όχι μόνο στοιχεία για το είδος του προβλήματος, τις διακρίσεις που υφίστανται, αλλά για όλα τα θέματα τα οποία καλύπτουμε στην έκθεσή μας, την οποία δεν μπορέσαμε να παρουσιάσουμε στο σύνολό της σήμερα, υπάρχουν στοιχεία τα, οποία λείπουν, δεν, υπάρχουν στοιχεία για, για ορισμένες ομάδες παιδιών, δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία σε ορισμένα κράτη μέλη αναπτύσσονται δίκτες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ε, ε, πολιτικές, σε άλλους ε, τομείς όπου γίνονται τακτικά έρευνες και μελέτες και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από αυτές τις πιο γενικευμένες πολιτικές. Αλλά Πολλέ πολλές φορές η κατάσταση για παιδιά με αναπηρίες δεν λαμβάνεται υπόψη βάσει συγκεκριμένων στοιχείων για τα παιδιά αυτά, αλλά βάσει στοιχείων που υπάρχουν σε γενικότερες μελέτες. Έχουμε ορίσει κριτήρια, ε, ε, τα οποία δεν παρουσιάσαμε σήμερα, αλλά τα βρίσκεται στο συμπέρασμα της έκθεσής μας. Αναγράφονται εκεί. Η έκθεσή μας περιλαμβάνει ένα μέρος ε, με όλες τις συστάσεις και σας καλούμε να μελετήσετε αυτό το ε, τελευταίο ε, τμήμα της μελέτης μας, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Πιστεύω, τώρα όσον αφορά το άλλο θέμα, το ότι δεν έχουμε δεν, τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, στην έκθεσή μας λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα για παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, εξαιρείται οποιαδήποτε δράση για τα παιδιά από το πεδίο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή, έχει αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση να χειριστεί το θέμα των διακρίσεων και της καταπολέμησης της επιβολής διακρίσεων σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό δεν αποκλείεται διόλου η δυνατότητα να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που δεν αναγράφεται ως συγκεκριμένη αρμοδιότητα αλλά αναγράφεται μόνο ως στόχος. Άρα λοιπόν δράσεις είναι δυνατόν να υπάρξουν. Όσον αφορά τώρα το θέμα της στέγασης, της ικανοποιητικής στέγασης, απαντώντας στην κυρία Γκυγιόμ, είναι σωστό ότι το θέμα αυτό της στέγατης συνδέεται με τις ε, διακρίσεις, ε, τις αρνητικές διακρίσεις. Όταν λέμε ε, ικανοποιητική στέγαση, reasonable accommodation, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα χρήσιμο μέσο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διευκολύνουμε τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες αλλά και ενηλίκων με αναπηρίες να στεγαστούν κατάλληλα. Είναι μία δύσκολη έννοια διότι υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα τα οποία ε, για τα οποία έκριναν ισπανικά δικαστήρια ότι χρειάζεται να παρέμβουν οι αρχές. Θα πρέπει ορισμένα από τα δικαιώματα αυτά να καλύπτονται από τι αρμόδιε αρχέ άσχετα από το κόστος. Άρα στο δικαστήριο δεν μπορεί κανεί να κάνει μία προσφυγή ή να προβάλλει το ε, απαιτήσει βάσει του, του, της ορολογίας εύλογο ή ικανοποιητικό ή επαρκές. Πρέπει να αρμηνεύσουμε ε, πιο συγκεκριμένα την ορολογία αυτή, τον όρο αυτή. Και εδώ ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή να ορίσουμε καλύτερα τι εννοούμε ακριβώς με αυτήν την ορολογία. Δεν είναι σαφής, είναι συγκεχημένη η έννοια αυτή όπως και η έννοια της ε, αναπηρίας των ειδικών αναγκών. Δεν είναι εναρμονισμένη η εμπειρία αυτή και θα πρέπει ε, να έχουμε καλύτερη, ε, καλύτερους ορισμούς για το ποσοστό, για τα ποσοστά αναπηρίες που, που πρέπει να εφαρμόζονται ή να κρίνονται στη μία στην άλλη περίπτωση για τα παιδιά αυτά. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα θέματα. Το άλλο θέμα της ανεργίας που τέθηκε δεν ε, κάναμε αυτήν την ε, διασύνδεση. Εμείς μελετήσαμε την, ε, την, το θέμα της παιδείας της εκπαίδευσης. Στη μελέτη μας, μία πτυχή την οποία, την οποία μας τόνισαν οι εμπειρογνώμονες, είναι η εξής. Μας είπαν ότι παρόλο που τα παιδιά με αναπηρίες έχουν ε, υψηλό, καλό, καλή μόρφωση, καλή εκπαίδευση στα σχολεία και πολλές φορές ε, στα λύκεια ή στο πανεπιστήμιο, επειδή είναι υποχρεωτικό να τους παρασχεθεί δηλαδή αυτή η παιδεία, ε, όταν ε, ολοκληρώσουν τη βασική τους παιδεία, ο ορισμός των παιδιών με αναπηρία που προχωρεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πέφτει δραματικά, είτε διότι ε, δεν έχουν τη δυνατότητα, είτε διότι δεν έχουν την αυτοπεποίθηση και τη βοήθεια να προχωρήσουν. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας. Άλλες ερωτήσεις. Εάν όχι, θα προχωρήσουμε στην ατζέντα μας. Προτού όμως ευχαριστήσω τις δύο εκπροσώπους ε, που παρουσίασαν ε, εκ μέρους της ομάδας αυτή την εξαιρετική μελέτη, ε, την κυρία Μέρενς και την κυρία Μπαλεστέρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες μου και θα προχωρήσουμε στο σημείο 5 της στο σημείο. 9. Ναι που είναι ο δικός χάρτης κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω γενετησίου προσανατολισμού και της ταυτότητας του φίλου. Η κυρία Λου, Λούνατσεκ είναι η συγγήτρια και το θέμα μας εδώ είναι ε, τι ε, πολιτική πρέπει να εφαρμόσουμε για να καταπολεμήσουμε ακριβώς ε, ο, τους, ε, τα άτομα αυτά ε, που υφίστανται ε, διακρίσεις λόγω του, του γενετής προσανατολισμού ή του φύλου. Θα ακούσουμε λοιπόν την εισηγήτρια και μετά θα ακούσουμε τους γεώδεις εισηγητές. Κυρία Λούνατσεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή που ήδη από την αρχή αποδέχθηκε να αναλάβουμε αυτήν την ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και επίσης που μου την εμπιστεύτηκε. Γιατί το ζήτημα είναι σημαντικό. Χτες το βράδυ στη Βιέννη, από που κατάγομαι, διοργανώνεται το φεστιβάλ κινηματογράφου Queer. Και ένα έργο που παρουσιάζεται η ιστορία ενός ε, άνδρα από την Πολωνία που έπεσε θύμα ομοφοβίας και βίας. Έχει αναγνωρίσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια αυτή η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδο στην καταπολέμηση της ομοφοβίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά πολλά απομένουν να γίνουν και αυτά προσπαθώ να αναδείξω με την έκθεσή μου. Επίση αυτή η έκθεση, αυτή η πρωτοβουλία δεν ε, έρχεται από το πουθενά, δεν ουρανοκοτεύεται γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια, όχι στην Επιτροπή Λίμπε, δέκα φορές στην Ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προετοιμάσει μια τέτοια χάρτα κατά πολέμηση της ομοφοβίας και να την παρουσιάσει, να την παρουσιάσει τα κράτη-μέλη σε εμάς. Ωστόσο η Επιτροπή αδράνησε και θεωρήσαμε εμείς ότι από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει νόημα να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία, να πιέσουμε ε, έτσι ώστε να υιοθετηθεί αυτός ο χάρτης, να εξηγήσουμε γιατί είναι απαραίτητος και να καταδείξουμε τι μπορεί να κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Το πρώτο θέμα, γιατί είναι απαραίτητος ένας τέτοιος χάρτης. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών δικαιωμάτων παρουσίασε το καλοκαίρι μια ε, στατιστική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 39.000 άτομα από όλα τα κρατημέλη και απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις. Τα στατιστικά αυτά νομίζω ότι μπορούν να, ε, ε, στα, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά για την έκθεσή μας. Το 1 τρίτο αυτών των των ομοφυλοφίλων, ε, μαθαίνουμε από αυτή την έκθεση, έπεσε θύμα διακρίσεων. Το 26% έχει δεχθεί επίθεση, απειλήθηκαν με βία. Το 35% μεταξύ των τρασεξουαλικών, μάλιστα, ε, έχει δεχθεί επίθεση ή ε, απειλήθηκε με βία. Παρά το γεγονό ότι απαγορεύονται διακρίσει στον χώρο τη εργασία, πολλοί από αυτά τα άτομα έχουν πέσει θύμα ε, τέτοιων διακρίσεων και μόνο το 10% αισθάνονται αρκετά ασφαλείς έτσι ώστε να καταγγείλουν τέτοιου τύπου διακρίσεις στην αστυνομία. Δείχνουν λοιπόν αυτοί οι αριθμοί ότι πολλά απομένουν να γίνουν. Πολλοί μερικές φορές φέρνουν το επιχείρημα μα δεν υπάρχει νομική βάση στην ε, συνθήκη για να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως υπάρχει το άρθρο 10 της συνθήκης που καθιστά σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση καταπολέμησης της, ε, των διακρίσεων όταν ε, καθορίζει και αναλαμβάνει δράση. Επίσης υπάρχουν και άλλες, άλλοι τομείς δραστηριότητες στους οποίους η Επιτροπή έχει προτείνει την καταπολέμηση των ε, διακρίσεων. Για παράδειγμα, την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω της αναπηρίας, για τους Ρωμά και για την ισότητα των δύο φύλων. Έχουμε τη στρατηγική για την απειρία, την στρατηγική για την ισότητα των ε, δύο φύλων. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων. Θεωρεί λοιπόν η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζω ότι ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο νομικό κείμενο που αναφέρεται στους ΛΟΑΤ. Κοντά στην παρουσίαση της έκθεσης της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 11 υπουργοί ε, αρμόδιοι για τα ζητήματα των διακρίσεων από τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την υποστήριξή τους για μια τέτοια, ε, ένα τέτοιο νομικό κείμενο για την καταπολέμηση των διακρίσεων των, κατά τον συγκεκριμένο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει υποστήριξη. Με την έκθεση που σας παρουσιάζω, εξηγώ γιατί χρειάζεται ένας τέτοιος χάρτης και, τι θα ε, προσφέρει. Με την έκθεση επίσης καλώ όλους τους αρμόδιους φορείς και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο των κρατών μελών να ξεκινήσουν να εργάζονται έτσι ώστε να ετοιμαστεί ένα προσχέδιο ένα τέτοιου οδικού χάρτη. στα έγγραφα που σας δίνει με η γραμματεία θα διαπιστώσετε ότι έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Οι εκθέσεις δεν πρέπει να είναι πολύ μακροσκελείς, γι' αυτό προφανώς δεν μπορούσαμε να βούμε σε όλες τις λεπτομέρειες και να εξηγήσουμε όλες τις δράσεις που θα θέλαμε να αναλάβουμε. Επομένως υποβάλλω ορισμένες τροπολογίες που αφορούν κυρίως τα εξής σε ποιους τομεί θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, ε, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία συνάθρηση, την υγεία, την εργασία, την ε, καταπολέμηση των διακρίσεων ε, όσον αφορά την πρόσβαση στα αγαθά και τι υπηρεσίες, τα δικαιώματα των πολιτών, το δικαίωμα μετακίνηση. Διάφορου τέτοιου τομεί. Τροπολογία σα την είχα αποστείλει και ηλεκτρονικά. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν ακούσουμε και από τους της εισηγητές. Πιστεύω ότι σε τέτοιου τύπου θέματα, τα οποία προκαλούν δυστυχώς ακόμα αντιδράσεις στην κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η αρχή της επικουρικότητας γίνεται πλήρως σεβαστή. Και ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να προτείνει θετικά παραδείγματα, παραδείγματα προς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την ίδια ή από κράτη-μέλη για να δείξει στα κράτη-μέλη περί τίνος πρόκειται αυτή η πρωτοβουλία και ευχαρίστως να συνεργαστώ ε, με όλους τους συναδέλφους, με όλους τους σκιώδους εισηγητές. Και ας μην ξεχνούμε ότι η αξία της ισότητας βρίσκεται στη βάση Τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω λοιπόν ότι θα υποστηρίξετε την εκθέσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λούνατσεκ. Τώρα ας περάσουμε στη συζήτηση. Ας έχουμε κατά νου ότι στις 11 ε, έχουμε και την ψηφοφορία. Να το έχετε λοιπόν αυτό κατά νου, επομένως ε, να είστε συνοπτικοί. Βοηθήστε μας με το χρόνο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μετσόλα, η οποία είναι σκιώδη εισηγήτρια για αυτό το ζήτημα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία και για όλη τη τη δουλειά για την έκθεση. Νομίζω ότι εν γέννη οδεύει προς το στην κατεύθυνση καθώς βασίζεται στο ψήφισμα το οποίο συμφωνήσαμε πέρσι. Όπως είπε και η κυρία Λούνατσεκ, πολλά έχουν γίνει, αλλά πιστεύω ότι πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίζουμε να καταπολεμούμε την εισαγωγή διακρίσεων κατά τον ε, ΛΟΑΤ και είμαι σίγουρη ότι η ευρεία συνένεση μπορεί να επιτευχθεί σε πολλούς τομείς και εγώ θα το διασφαλίσω μαζί με την ομάδα μου. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις σε ορισμένα σημεία. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες όπου περιλαμβάνονται προτάσεις που μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω. Γιατί ενώ συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα αυτά τα ζητήματα, εγώ θέλω να διασφαλίσω, έχοντα κατά νου και όσο είπε η κυρία Λούλτσο και για την επικουρικότητα, ότι το κείμενο είναι πολύ σαφές και δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να νομοθετήσουν σε αυτόν τον τομέα, σε κάποια άλλα σημεία. Είναι πάρα πολύ καλή διατύπωση, αλλά μπορεί να είναι κάπως δύσκολο να λειτουργήσουν στην πράξη λόγω γραφειοκρατίας και ε, νομίζω ότι σε κάποια άλλα σημεία πάμε πολύ μακριά στο θέμα των θετικών διακρίσεων και πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Πάντως η αρχική μου αντίδραση είναι θετική και νομίζω ότι αν ε, όλοι έχουν ε, τη διάθεση να συμβιβαστούν θα, θα καταλήξουμε με ένα κείμενο που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μετσόλα. Και ο, Μισελ, ο κύριος Μισελ εκπροσωπεί την κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ εξ ονόματο ε, της ομάδας ε, των φιλελευθέρων. Ε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Σοφή Ιντβελτ που δεν μπορεί δυστυχώ να είναι εδώ και ξέρετε πόσο πολύ την ενδιαφέρουν όλα αυτά τα ζητήματα. Επίση, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λούνετσα για την εκθεσή τη. Ε, φυσικά έχει την πλήρη υποστήριξη τη ομάδα των φιλελευθέρων. Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετική η έκθεση. Θέλω να υπονθυμίσω ότι η πρόταση για ένα χάρτη πορεία προέρχεται από την κυρία Ιντβελτ και από την ομάδα Άλντε. Εμείς ε, επιμείναμε για τη μελέτη για τον οδικό χάρτη και για την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που πετύχαμε το στόχο. Τώρα, ως σκιώδης ε, εισηγητής έχω συμπεριλάβει και τα θέματα των ανθρώπων ΛΟΑΔ ε, στην εκθεσή μου. Έτσι λοιπόν και πάλι συγχαίρω την κυρία Λούνατσεκ και τον κύριο Κάτσμαν και όλους όσους εργάζονται για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών χωρίς καμία εξαίρεση. Ευχαριστώ κύριε Μισελ κυρία Ένστ. Ähm, Ευχαριστώ. Ο σκιώδης συζηγητής ε, σε εμάς είναι ο κύριος Γιόγκ και θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας να πω τα εξή. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που υπάρχει αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, ε, έχει αργήσει αρκετά, έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα. Είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε αυτήν την έτσι το φαινόμενο της ομοφοβίας και της βίας γίνεται όλο και πιο απειλητικό και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε η εμπειρία της ε, στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρωμά μας δείχνει ότι πρέπει να καταλήξουμε σε πολύ συγκεκριμένε συμφωνίες γιατί ξέρουμε ότι είναι εκτός του κοινοτικού δικαίου. Όμως πρέπει να υπάρχουν υποχρεώσεις των κρατών μελών, πρέπει να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να τηρούν ορισμένα πράγματα και είναι πολύ σημαντικό αυτό και η Κομισιόν θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί και θέλει να χειριστεί παρόμοια θέματα. Είχαμε μία συζήτηση στο παρελθόν παρόμοια και τελικά τίποτα δεν έγινε σε σχέση με τους Ρωμά. Τώρα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση γιατί με ανισχούν ιδιαίτερα τα, οι συστάσεις αν θα είναι υποχρεωτικές, δηλαδή το θέμα της υποχρεωτικής ε, εφαρμογής. Δεύτερον, θα παρακαλούσα να λάβετε υπόψη μία άλλη ε, πτυχή επί της οποίας υποβάλλουμε μία τροπολογία. Ε, όταν μιλούμε για το Β, Γ, Δ, δηλαδή τα πράγματα τα οποία θέλουμε να εφαρμοστούν, ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη το, το φύλλο, ε, την ταυτότητα του φύλου. Επίσης, το ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Μην το χάσουμε και αυτό από, τα, από τον ορίζοντά μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα μέσα ενημέρωσης, διότι και αυτά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο είτε θετικά είτε αρνητικά στο όλο θέμα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματιέ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρουνατζέκ για την έκθεση που μας παρουσιάζει. Είναι μια πολύ καλή έκθεση. Δεν έχω δει τις τροπολογίες, αλλά φαντάζομαι ότι συνάδουν με την έκθεση, η οποία καλεί σε έναν απαραίτητο χαρτί πορείας. Νομίζω ότι είναι η δέκατη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας που εξετάζουμε αυτό το ζήτημα και ο σκοταδισμός της Κομισιόν πραγματικά είναι ανησυχητικό, κυρίως όταν ξέρουμε ότι 10 κρατημέλη και 11 υπουργοί εξέτασαν αυτό το ζήτημα και επομένω είναι πολύ καλό που το Κοινοβούλιο επανέρχεται στο τέλος της θητείας. Και καλό κουράγιο κυρία Λούναξε και στους Κιώδης και φαντάζομαι ότι η ομάδα μας ε, θα υπερψηφίσει την έκθεση αυτή και όλοι θα συμφωνούν. Ευχαριστώ, κύριος Μωράης. Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρους του κυρίου Κάσμαν, ο οποίος ε, έχει εμπλεκεί τα μάλα στην έκθεση αυτή. Η κυρία Λούνατσεκ παρουσίασε μια έκθεση και νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται εδώ ακριβώς η ανάγκη για μία απάντηση και για ένα οδικό χάρτη που το χρειαζόμαστε απαραίτητα. Νομίζω ότι υπάρχουν διδάγματα που προκύπτουν από αυτή την έκθεση, καθώς μιλάμε για το θέμα των Ρωμά. Παραδείγματο χάρη η νομική βάση υπάρχει για την εισαγωγή διακρίσεων, αλλά η εφαρμογή ε, είναι πολύ αδύναμη ανεπαρκής και άκουσα κάποιους συναδέλφους εδώ να μιλούν ε, για την επικουρικότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεως στα κατά και τις Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονιστεί στην έκθεση και πρέπει να είμαστε σαφείς ότι οι Υπουργοί Ισότητας ε, θα ε, πρέπει να συμφωνούμε με την έκθεση αυτή και πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Θα χρειαστεί λοιπόν η κυρία τσεκ την υποστήριξή μας. Δεν είναι καλοπιστική έκθεση αυτή, πρέπει να την υποστηρίξουμε πολιτικά. Νομίζω ότι είναι πλήρης η έκθεση και η ομάδα ε, που ανταποκρίθηκε μας ε, έχει δείξει ότι υποστηρίζει και το ίδιο ισχύει και από τον κύριο Κάσμαν. Δεν μέγιστη υποστήριξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μωράης που εκπροσωπεί τον κύριο Κάσμαν Νομίζω ότι ο κύριος Μπρόγκς έχει ζητήσει το λόγο. Yes. <coughs> People of... Μάλιστα. Άνθρωποι όλων των ε, πεπιθήσεων και προτιμήσεων ε, δεν θα πρέπει να είναι σήματα κακοποιήσεων και καταχρήσεων. Ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την επαγγελματική τους δραστηριότητα και την εισοδηματική τους πηγή. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την ομοφοβία που γεωλεκτικά σημαίνει την, το φόβο του ιδίου, του, του, του παρομοίου στοιχείου διαπιστώνουμε μία έλλειξη σεβασμού και μία εχθρότητα στη συμπεριφορά η οποία δεν είναι ανεκτή και πρέπει να αλλάξει. Δεν θα πρέπει μία κρατική αρχή ή μία υπερκρατική αρχή να επιβάλλει την αλλαγή της συμπεριφορά. Το κράτος θα πρέπει να αποθαρρύνει τη βία και βια η συμπεριφορά. Ε, έχουμε συζητήσει το θέμα και στο παρελθόν, αλλά και ακόμα το Βατικανό έχουμε διαπιστώσει ότι ε, εφήρμοσε μία ρητορική μίσους και μία σχετική αρνητική πολιτική. Ε, θα, θα πρέπει λοιπόν ε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τα Ιερά Βιβλία, από τις βίβλους, ορισμένα αποφθέγματα και παραγράφους τις οποίες τα άτομα αυτά τα, βρίσκουν, τα θεωρούν προσβλητικά, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά ο γενετήσιος προσανατολισμός και τα άλλα στοιχεία που καθορίζουν έναν άνθρωπο ε, είναι προσωπικά, είναι ατομικά και το θέμα είναι ότι δεν υποχρεώνουν υποχρεώνεται καθένας να ανακοινώνει ποιες είναι οι προτιμήσεις του. Αλλά αυτό το οποίο είναι υποχρεωτικό του νόμου είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της συμπεριφοράς, προσωπικής ζωής. Ε, και πολλά, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ακριβώς αυτό το δικαίωμα της ε, ελεύθερης έκφρασης. Παρόλο, τώρα ε, διαπιστώνουμε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταργούν και απαγορεύουν την ελεύθερη έκφραση και κυνηγούν αυτούς που την εκφράζουν. Ο πρόεδρος, Ωραία. Αφού ακούσαμε λοιπόν την συγγήτρια και τους Κιώδης, θα ακούσουμε την ε, Κομισιόν. Καλημέρα σας. Ε, Είμαι, εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και εργάζομαι στη, στο τμήμα κατά των διακρίσεων, κατά πολέμηση των διακρίσεων. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια, ε, διότι και εμείς συμμεριζόμαστε τις, ε, τους φόβους και τις ανησυχίες της και ε, είμαστε υπέρμαχοι της καταπολέμησης των διακρίσεων. Είναι πολύ δύσκολο για μας να εκφράσουμε

στοιχεία τα οποία αποτελούν μέρος της συζήτησης. Το πρώτο είναι ότι η Κομισιόν τώρα ε, ε, σε λίγο θα συμπληρώσει, θα ολοκληρώσει την εντολή της και μπορεί να ανανεωθεί τον Μάρτιο. Ε, we are looking into the future now. So... συγγνώμη, η έκθεση θα ψηφιστεί το Μάρτιο στο Κοινοβούλιο και Εμείς ε, θα διαμορφώσουμε την πολιτική μας ε, για το επόμενο έτος και το θέμα της, ε, της μεταχείρισης και της πολιτικής μας για τα άτομα, για τους ΛΟΑΤ αποτελεί μέρος της γενικής μας προσέγγισης. Το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης ξεπερνάει την, ε, τις πολιτικές ε, δηλώσεις, την, την πολιτική μας ε, θέση, αλλά όπως σας είπα δεν είμαι εξουσιοδοτημένος, ούτε μπορώ σήμερα να εκφράσω τη θέση μου. Τη θέση της Επιτροπής δηλαδή. Και τέλος, όπως ανέφεραν πολλά κράτη-μέλη, το θέμα του καταμερισμού της ευθύνης δεν είναι μόνο η Κομισιόν η οποία θα πρέπει να ενεργήσει εδώ, αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να παίξουν το ρόλο τους, πρέπει να σεβαστούμε την, την αρχή της επικουρικότητας και από πολιτικής απόψεω πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τα δεκα, ε, όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο τα 11 που είναι πρόθυμα να ακολουθήσουν μια στρατηγική, αλλά και τα υπόλοιπα 17. Ε, διότι ε, διαφορετικά θα, πρέπει να εκδώσουμε μία λευκή βίβλο η οποία να ε, δώσει μία βίβλο η οποία θα ορίζει το, το μήνυμα και το πνεύμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς θέλουμε να συμπαρασύρουμε την πλειοψηφία των κρατών μελών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι με το μέρος μας, η κοινωνία των πολιτών είναι ε, και θέλουμε τώρα να καταφέρουμε να έχουμε μια εύλογη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ που, έχετε διατηρήσει αυτό το πολύ σημαντικό θέμα στην ατζέντα σας. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε την Κομισιόν, τώρα δίνω το λόγο στην συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω. Ο Πρόεδρος ε, ζητώ όσοι έρχονται στην αίθουσα να το κάνουν ήσυχα γιατί προσπαθούμε να ακούσουμε την εισηγήτρια. κυρία Λούνατσεκ. Ωραία, ξαναρχίζω. Ε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο σχόλιο που έκανε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Δηλαδή αυτό που είπατε ότι ήδη έχει εκφραστεί υποστήριξη για την κατάκτηση ενός τέτοιου τύπου ε, στρατηγικής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από ορισμένα κρατημέλη, από την κοινωνία των πολιτών. Σίγουρα αυτό που λείπει είναι να πείσουμε τα υπόλοιπα κρατημέλη και ελπίζω να συνεργαστούμε και να το πετύχουμε αυτό. Αποδέχομαι ότι προφανώς δεν μπορείτε να εκφέρετε γνώμη ακόμα, αλλά είμαι βέβαιη ότι η τρέχουσα επιτροπή και η επόμενη επιτροπή θα την εξετάσουν προσεκτικά την έκθεση ίδιας πρωτοβουλία που προετοιμάζει το Κοινοβούλιο και θα υπάρξει σωστή συνεργασία. Να ευχαριστήσω επίσης τους κοιόδης ή τους εκπροσώπους τους. Με χαρά διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη ε, πρώτα απ' όλα για το να αναλάβουμε αυτήν την πρωτοβουλία και δεύτερον για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης σε μεγάλο βαθμό. Επίσης θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδελφούς ότι η επικουρικότητα είναι ε, σημαντική και για εμένα, αλλά πρέπει να εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της επικουρικότητας. Ε, συνάδελφος αναφέρθηκε στο να εισάγουμε και την οπτική του φίλου για παράδειγμα να αναφερθούμε στα ιδιαίτερα προβλήματα των λεσβιών ή επίση και το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωση. Θέλω να επιμείνω σε αυτό, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωση να αναφέρονται ε, στου ομοφυλόφιλου και στι λεσβείε και στα άτομα αυτά μόνο όταν υπάρχουν προβλήματα και ποτέ όταν η κατάσταση είναι φυσιολογική και νομίζω αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ένα μικρό σχόλιο για τον συνάδελφο τον κύριο Μπρόν. Εδώ δεν μιλούμε για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Μιλάμε για την εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από αυτές τις θεμελιώδεις αξίες είναι η ισότητα και το δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που καθιερώνονται στι συνθήκε. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω του σκιώδει εισηγητέ που εξέφρασαν όλε αυτέ τι απόψει, να ε, ευχαριστήσω επίση το προσωπικό τη ομάδα μου και τη γραμματεία για την υποστήριξη. Προσβλέπω στη συνεργασία μα έτσι ώστε να καταρτήσουμε ένα χάρτη, μια χάρτα η οποία θα δείξει και στην κοινότητα των ΛΟΑΤ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να φτιάξει ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να ζουν χωρίς φόβο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για όλα αυτά, για την έκθεση, για τις παρατηρήσεις σας. Θα σταματήσουμε τη σχετική συζήτηση εδώ. Να σας υπενθυμίσω της ε, προθεσμίας. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 18η Νοεμβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ωραία. Ενημέρωσα λοιπόν και για την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών και ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το σημείο 9. Δεν έχουμε καθυστερήσει καθόλου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ακριβώς την ώρα της στην ψηφοφορία. Σα ζητώ να είστε συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Πρώτα απ' όλα ε, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική σας κάρτα. Όσοι δεν έχετε φέρει την ηλεκτρονική κάρτα, ε, παρακαλώ να μας, το, να μας ενημερώσετε για να μπορέσουμε να καταμετρήσουμε σωστά τις ψήφους. Ναι, όσοι δεν έχουν κάρτα να μας το πούν. Για να υπολογίσουμε και την απαρτία και την κατανομή των ψήφων. Κυρία Ζντάνοκα, δεν έχετε ε, κάρτα, επομένως θα σηκώνετε το χέρι σας. Το ίδιο ο κύριος Ρομέρο. Υπάρχει κάποιος άλλος που δεν έχει κάρτα. Ε, θεωρώ ότι οι υπόλοιποι είστε έτοιμοι. Έχει διανεμηθεί ο κατάλογος φορείας σε όλες τις ομάδες. Έχουμε ψηφοφορία για την επόμενη μισή ώρα. Είναι το σημείο 10 τη ημερήσια διάταξη. Προποθέσει εισόδου και διαμονή επικών τριών χωρών με σκοπό την έρευνα, σπουδέ, αλλαγή μαθητών, έμιστη, ή άμιστη πρακτική άσκηση, ενθελοντική εργασία και την απασχόληση ω ε, βοηθών ΟΠΕΧ. Η εισηγήτρια είναι η συνάδελφο Σιλία Βίξτρο. Έχουμε λοιπόν την έκθεσή τη σε σχέση με αυτήν την ε, οδηγία που αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία. Κυρία Βίξτρομ, δεν θέλετε το λόγο. Επίση θα ψηφίσουμε και για την εντολή διαπραγμάτευση. Ξεκινούμε λοιπόν με την ψηφοφορία επί τη έκθεση. Λοιπόν, Γιούρι 2, υπέρ, κατά, απο, απορρίπτεται. Α, αποχές, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, ξέχασα. <laughs> Απορρίπτεται. Έμπλ 13. Εδώ έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος, υπέρ. Those against. Abstentions. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία, το 66 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, ο πρόεδρος είπε 16, αλλά δεν πειράζει. Η 66 είναι. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε η ψηφοφορία... 15 έναντι 33 απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 68 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 69 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Τέσσερα. Α, όχι. οι πέντε υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Δεκαπέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εμπλ 16. Σε δύο τμήματα. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο μέρος. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εμπλουά 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 72 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, Ξανά την 71 παρακαλώ, υπέρ. Α, ε, έγινε ηλεκτρονικός έλεγχος. 4 έναντι 31. Απορρίπτεται. Υπέ, ε, το 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Employ 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Employ 23 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Α, αυτή ήταν 24. απορρίφθηκε 24. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εμπλό 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79. Υπέρ κατά, αποχές, δεκτή, 27 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 28, δύο, δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπο... Τροπολογία 8, 80, 81, ταυτόσημες, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 29. έχει, έχει καταπέσει. Καταπίπτει. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά εποχές ε, εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή Οπολογία 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 6, ε, ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε στην employ 41, υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτή. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπάρχει Ξεχωριστή ψηφοφορία, πως τη ζήτησε το ΕΛΚ. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Employ 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 114. Καταπίπτει. Αχα, προχωρούμε λοιπόν στην συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά άποχες. Δεκτή. 150. Πάμε στην 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή α, η 50 κατά πίπτη η 31 31 ισχύει δεν καταπίπτει ψηφίζουμε την 31 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δε, δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33. Α, ένα λεπτό. 150. Η 153 έγινε δεκτή. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 153. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Προχωράμε στην 155 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος 155 παρακαλώ. 155 ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. Ε, δεκτή. 26-24. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 157 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, συμβαστική 11 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο μέρος συμβαστικής 11 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 162 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 63, 163 και εμπλόι 52, ταυτόσημες, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Αμφότερες, 37, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 38, γλωσσική, δεν έχουμε πρόβλημα, 39, υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Employ 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 41. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 42. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 43. κλωστική, Προχωρούμε. Employ 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Employ 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 13 δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο μέρος υπέρ κατά, αποχές, δεκτό. Employ 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ κατά, αποχές, δεκτή, employ 10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 61, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 2, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 62 παρακαλώ. Ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 63. Από ό,τι φαίνεται, είναι, είναι η τροπολογία 2 που δεν είναι σίγουρη η έκβαση ο πρόεδρος, μπορούμε παρακαλώ να επανέλθουμε στην τροπολογία 2 και να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Απορρίπτεται. Έτσι δεν είπα. Ναι. Ωραία. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κα, κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Ψηφίζουμε το κείμενο ως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικός έλεγχος του τροποποιημένου κειμένου. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 48 υπέρ. Μία αποχή, τρεις ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια Α, 49, 49. Μάλιστα. Συγχαρητήρια κύριε Βίξτρομ. 49 με, την, με τις ψήφους ε, διανατάσεως χειρός. Ωραία, ένα λεπτό. Τώρα ψηφίζουμε την εντολή, ψηφίζουμε την εντολή έναρξης ε, διαβουλεύσεων. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. 48, 49, υπέρ, μία ψήφος κατά και καμία αποχή. Ωραία. Τώρα κύριε Μπίξτον μπορείτε να μιλήσετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συμβολή τους. είναι η, ο τελευταίος μήνας αυτός για την εντολή και ήταν δύσκολο να συγκεράσουμε όλες τις απόψεις της ομάδας αλλά τα καταφέραμε και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Μαρία από τη Γραμματεία η οποία λάμπει είναι ένα στέρι και ευχαριστώ και όλους τους ε, συμβούλους, τους εμπειρογνώμονες, τους σκιώδους εισηγητές. Ε, συνεργάστηκα μαζί τους με μεγάλη χαρά. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα είναι λίγο ωφέλιμη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευχαριστώ όλους ε, όσους συνέβαλαν. for credit Ευχαριστώ κύριε Βίξτρομ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τη γραμματεία. Μπορείτε να αποχωρήσετε από την αίθουσα, αλλά ήσυχα. <laughs> Okay? If I have your attention. Ωραία. Να έχω την προσοχή σας και πάλι. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης σήμερα το πρωί. Το θέμα είναι η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος Ρόνι Σάρα Λάτφορτ. Να σας θυμίσω ποιο είναι το πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Αναφ... ε, υιοθετήθηκε το πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης το 2002. Ήταν μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που ελήφθη ποτέ στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικέ υποθέσεις. Έχει ε, αλλάξει ε, ε, δραματικά την κατάσταση. Το παλαιότερο σύστημα για τις παραδόσεις κρατουμένων ήταν πολύ ε, γραφειοκρατικό και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, το βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό. Ωστόσο, έχει έρθει η στιγμή να αναθεωρηθεί αυτό το σύστημα και θα ακούσουμε την, την παρουσίαση από την εισηγήτρια την κυρία Λάτσφορτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε κι εσείς, Πρόκειται για έκθεση ίδια πρωτοβουλία επί νομοθετικού ζητήματο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Με χαρά ανέλαβα αυτή την, αυτό το έργο και να ευχαριστήσω και τους σκιώδες συζητητέ με τους οποίου έχουμε συνεργαστεί και κατά το παρελθόν ε, σε ζητήματα συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις. Μάλλον έχουμε γίνει παρεάκι. Έχω ασχοληθεί με ζητήματα αυτά Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ήμουν εισηγήτρια για τον ε, πρώτο δικό χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα, την ε, εφαρμογή τους στις ε, ποινικέ υποθέσεις. Πάντα με ενδιαφέρε το ζήτημα της, του Ευρωπαϊκού Εντέλματος Σύλληψης. Συμμετέχω επίσης και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα ή έχω ασχοληθεί προσωπικά και με ατομικές υποθέσεις. Είχαμε δύο συναντήσεις με τους ε, σκιώδες μέχρι τώρα και μια δημοσία ακρόαση στην Άλντε πριν λίγες εβδομάδες που νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη. Η τρίτη συνάντηση των σκιωδών θα γίνει αύριο. Για ε, γνωμοδοτήσεις ιδίας πρωτοβουλίας σαν και αυτήν, κάτι που είναι καινούριο με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, δίνεται η δυνατότητα στον εισηγητή να κάνει μια προφηταρχική εξέταση και να αξιοποιήσει τη συνεισφορά δύο ε, ειδικών. Οι δύο εμπειρογνώμονες λοιπόν που θα κάνουν αυτή τη μελέτη είναι η κυρία Άναν Ντούμπε, ειδικό σε ζητήματα εκδόσεων ε, και γενικότερα ε, ποινικού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και η καθηγήτρια προ, Αν ε, Βέμπερκ από το ELB, το Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, επίσης συντονίστρια του έκρε του Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Δικτύου για ζητήματα ποινικού δικαίου. Αυτοί οι δύο εμπειρογνώμονε λοιπόν, εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν τα προκρατικά αποτελέσματα της μελέτης που διεξάγουν αύριο. Όπως είπατε, ο στόχος του της απόφασης πλαισίου για το Ευρωπαϊκό ε, Ένταλμα Σύλληψης το 2002 ήταν να διευκολύνει την έκδοση ε, εγκληματιών και να ε, διασφαλίσει ότι αυτά τα άτομα θα προσάγονται στην δικαιοσύνη, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία και το χρονοβόρο παλαιότερο σύστημα εκδόσεων που είχαμε, μέσω της ε, αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών ε, αποφάσεων και βελτιώνοντας την συνεργασία. Το Ευρωπαϊκό Εντέλμα ε, σύλληψη λοιπόν διευκολύνει τις εκδόσεις πολιτών μεταξύ κρατών θέτοντας αυστηρά χρονικά περιθώρια και καταγράφοντας επακριβώς με βάση ποιους λόγους μπορεί ένα κράτος μέλος να αρνηθεί μια τέτοια έκδοση και διάφορα άλλα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι το γεγονός ότι έχουμε ανοιχτά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αξιοποιείται από εγκληματίε. Παράδοση ε, υπόπτων επίσης πρέπει να διασφαλίζει το γεγονός ότι αυτά τα άτομα δεν θα κρατούνται ε, πέρα μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηταμένα αναμένοντας την έκδοσή τους και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει έχουν παρουσιαστεί κάποια προβλήματα στον τρόπο εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και κυρίως της ε, αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων. Κάποια από αυτά τα προβλήματα έχουν προκύψει από κακή ε, μεταγραφή της ε, νομοθεσίας, δηλαδή διαφορές μεταξύ του δικαίου των κρατών μελών. Αυτό ίσως θα μπορούσε να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα μέσω δράσεων που θα αναλάβει το 2016 η Επιτροπή ενώπιον του δικαστηρίου. Διάφορα ζητήματα τα ανακύπτουν. Να σας αναφέρω μερικά. Τα ευρωπαϊκά εντάλματα έχουν ένα χρονικό περιθώριο που όπως είπα είναι πολύ σημαντικό για να μην υπάρχει κράτηση επί ε, μεγάλο χρονικό διάστημα προφυλάκηση επί μεγάλο χρονικό διάστημα και επίσης να είναι ε, γρήγορο το, η, η, εφαρμογή του συστήματος. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη συχνά δεν σέβονται αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Επίσης δεν προβλέπονται καθόλου χρονικά, το, δεν προβλέπεται καθόλου ένα χρονικό πλαίσιο, ένα όριο χρονικό για την μετάφραση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης και αυτό είναι ένα νομικό κενό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι το κράτος μέλος που έχει εκδώσει το ευρωπαϊκό Έντελμα σύλληψης έχει την υποχρέωση να αφαιρέσει οποιοδήποτε χρόνο προφυλάκησης δι, ε, δι, ε, ε, βρισκόταν υποκράτηση ο κρατούμενος σε οποιοδήποτε άλλος κράτος μέλος. Αυτό ήταν σημαντικό όσον αφορά την εναρμόνιση. Πρέπει το κράτος μέλος που τελικά στο οποίο τελικά παραδίδεται ο κρατούμενος, να λάβει υπόψη του το χρόνο προφυλάκησης που εξέτησε στα άλλα κράτη. Όμως αυτό στην πράξη δεν συμβαίνει. Και ο χρόνος προφυλάκησης ε, στο κράτος μέλος που εκτέλεσε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης πολύ συχνά αγνοείται. Και αυτό είναι πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζει η απόφαση πλαίσιο. Αυτά είναι κάποια από τα προβλήματα που θα έβαζα υπό τον τίτλο της μη εφαρμογής, μη σωστής εφαρμογής. Ένα άλλο κεφάλαιο προβλημάτων είναι αυτά που προκύπτουν από κενά για στο... ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, τα χρονικά όρια ε, δεν είναι σαφές εάν συμπεριλαμβάνουν τα... τις διαδικασίες έφεσης. οι να δεν αναφέρονται καν η άσκηση ειδικών μέσων. Επίσης το ζήτημα του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει, βρίσκεται στην καρδιά αυτής της προσέγγισης. Και το άρθρο 3 της απόφασης πλαίσιο αναφέρεται στην υποχρέωση των κρατών μελών να ε, σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Ωστόσο, κάποια ε, εθνικά δικαστήρια δεν έχουν φανεί πρόθυμα να δεχτούν να μην εκτελέσουν ένα ευρωπαϊκό ε, ένταλμα όταν υπάρχει ο κίνδυνο να μην γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επειδή αυτά δεν αναφέρονται ρητά ω λόγο απόρριψη αιτήματο στην απόφαση πλαίσιο. αλλά έχουμε περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι εξόφθαλμη η πιθανότητα ο κρατούμενος να μην έχει έντιμη δίκη. Και νομίζω ότι αυτό δεν ε, είναι ορθό, δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχυρίζεται ότι έχει οικοδομηθεί στα, ε, στη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έπρεπε να έχουμε έναν μηχανισμό που να εξασφαλίζει υψηλότερα ε, πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα έρευνα, Έρευνας, το οποίο αναφέρεται σε ε, ε, έρευνες που διεξάγονται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, όχι σε εκδόσεις κρατουμένων. Και σε αυτήν την διαπραγμάτευση έχουμε εισάγει ρητά μια αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή θα μπορεί ένα κράτος μέλος να απορρίπτει την εκτέλεση ενός τέτοιου εντάλματος όταν υπάρχουν και αναφέρω ε, εύλογες ανησυχίες ότι η εκτέλεση αυτού του εντάλματος θα αντίκειται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, για την, και στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν το κείμενο έχει συμφωνηθεί για το ένταλμα έρευνας, θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και για το ένταλμα ε, έκδοσης. Επίσης το ζήτημα της παροχής περαιτέρω πληροφοριών, εάν η εκτελούσα αρχή το ζητήσει, δεν προβλέπεται τέτοιο δικαίωμα όμως για το κράτος μέλος που έχει εκδώσει το έντελμα. Η Επιτροπή διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και διμερός και πολυμερός, αλλά από ό,τι, καταλα... έχω αντιληφθεί αυτό γίνεται κυρίως σε επίπεδο εισαγγελέων. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να ορίσουμε συντονιστέ στα κράτη-μέλη, στους οποίους θα μπορούσαν να απευθύνονται ερωτήσεις ε, που αφορούν το νομικό πλαίσιο θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει ένα ε, πρόγραμμα για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, Σύλληψης. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι το γεγονό ότι δεν υπάρχει μία συστηματική αναθεώρηση των σημάτων που βρίσκονται στο σύστημα Schengen, το οποίο οδηγεί πολλές φορές σε ε, συλλήψεις ε, χωρίς λόγο. Δεν είναι σαφές ποια είναι η σχέση του Ευρωπαϊκού Ένταλματο σύλληψης με αυτά τα σήματα Σέγγεν ή επίσης το τι συμβαίνει σε περίπτωση που ε, απορριφθεί ένα Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, σύλληψης από την εκτελούσα αρχή που σημαίνει ότι ο εν λόγω άνθρωπος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει γιατί θα παραμένει μέσα στο σύστημα Σέγγεν ένα σήμα που τον αφορά. Υπάρχει μια εξαιρετικά προβεβλημένη υπόθεση που συνέβη κάτι τέτοιο και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ε, συμφωνήσει ότι υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των ενταλμάτων, θα πρέπει να υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση των απορρίψεων των ενταλμάτων. Να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη υποτίθεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο τη ε, διαδικασία διερεύνηση ε, μια ποινική υπόθεση. Αλλά δεν είναι σαφή δεν έχει οριστεί σαφώς τι σημαίνει ακριβώς διερεύνηση μιας ποινική υπόθεσης. Ορισμένοι ισχυρίζονται ενώ άλλοι δεν συμφωνούν ότι πολλές φορές γίνεται κατάχρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης προκειμένου στην πραγματικότητα να προσαχθούν μάρτυρες ή για να γίνει μια ανάκριση στην προδικασία. Κάτι που δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο λόγος που δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Ελπίζουμε ότι βέβαια το Ευρωπα... η οδηγία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ή πιθανόν στο πλαίσιο της, του, του, Συμφώνου για την Αμοιβαία Δικαστική Συνεργασία στην Προδικασία να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία για να το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Υπάρχει επίσης ανησυχία για την δυσανάλογη χρήση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης, το οποίο εν μέρη προκύπτει από τις ε, διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων και στο δικονομικό επίπεδο και στο ουσιαστικό επίπεδο. Ένας εκπρόσωπος του Πολωνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης μας έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τα τροποποιήσεις στο Σύνταγμα και στην ομοθεσία της χώρας που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Πολωνία είναι παράδειγμα προς μίμηση σε αυτόν τον τομέα γιατί πολλά ε, ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης έχουν ε, απευθυνθεί προς τη χώρα αυτή. Έχει μια πολύ αυστηρή, ένα πολύ αυστηρό ορισμό του κατά πόσον το ένταλμα είναι σύνομο του κατά πόσον εξυπηρετεί το, τη, το, τη δικαιοσύνη, την απόδοση δικαιοσύνη. Γιατί έω τώρα η Πολωνία απέριπτε πολλά ευρωπαϊκά ανταλλήματα σύλληψης. Η Επιτροπή έχει αναφερθεί σε αυτό το θέμα στην εκθεσή της για την ε, υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ανταλλήματος Σύλληψης το 2011. Φαίνεται λοιπόν πως κάτι γίνεται. Ίσως όχι αρκετό όμως. Να μην είναι. Να αναφέρω επίσης ότι στην οδηγία για την Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας ε, καταφέραμε να συμφωνήσουμε και με το Συμβούλιο να υπάρχει ρητή αναφορά σε, μια αυστηρή, σε ένα αυστηρό έλεγχο της αναλογικότητας. Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί προηγούμενο για όλα τα ε, για όλη την νομοθεσία στη δικατιστική συνεργασία. Το Ρωμαίο Βασίλειο και άλλα κράτη-μέλη γνωρίζω <clears throat> ότι έχουν αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για να υπάρχει ο έλεγχος της αναλογικότητας πριν την εκτέλεση τέτοιων ενταλμάτων. Ίσως η Επιτροπή να θεωρήσει ότι αυτό αντίκειται στην απόφαση πλαίσιο, αλλά συμβαίνει. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από, έχουν προκύψει από το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα σύλληψης γιατί η διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκε ο κοινό χώρος δικαιοσύνης ήταν κάπως κατακαιρματισμένη. Ποινική συνεργασία. Από το 2011 που ασχοληθήκαμε με τα ζητήματα της κράτησης και της προδικασίας, δεν έχει υπάρξει νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι προφυλακισμένοι για μακρά χρονικά διαστήματα απλώς περιμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσης τους, ε, πολύ συχνά σε κακές συνθήκες κράτησης. Και τώρα παρατηρούμε ότι εθνικά δικαστήρια αρνούνται να εκτελέσουν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψη ε, ε, επιχειρηματολογώντα επί τη βάση των κακών συνθηκών κράτηση που θα αντιμετωπίσει ο κρατούμενο. Ε, υπάρχει μια τέτοια υπόθεση στην Ιρλανδία. Αυτό δημιουργεί λοιπόν πολλά προβλήματα. Μίλησε λοιπόν πριν για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο γενικά για την ποινική δικαιοσύνη, ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα αλλά δεν έχουμε κάποιο αντίστοιχο δίκτυο συνεργασίας των δικηγόρων υπεράσπισης. Αν και υπάρχουν ε, ανεπίσημα δίκτυα τα οποία υποστηρίζει χρηματικά η Επιτροπή, αλλά θεσμοθετημένα δεν υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο για να υποστηρίξει και να παρέχει εκπαίδευση στους ε, μαχόμενους δικηγόρους που υπερασπίζονται κρατουμένου. Και τέλος έχουν υπάρξει υποθέσεις όπου απλούστατα ε, συνελήφθησαν λάθος άτομα και κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν την πρωτοφανή κακοδικία. Ελπίζω ότι θα αναλυθεί μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να αναλάβει την ευθύνη και να αποζημιωθούν τα θύματα αυτών των περιστατικών. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα έχω καταγράψει. Ορισμένα από αυτά, όπως σας είπα, θα αντιμετωπιστούν από την άσκηση των ε, αρμοδιοτήτων ε, εφαρμογής της Επιτροπής, αλλά ε, τα συμπεριλαμβάνουμε σε άλλες οδηγίες, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα νομικής αρρωγής, Υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία κάπως θα μειώσουν τον πειρασμό που έχουν οι δικαστικές διοπτικές αρχές να καταχρώνται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Προφανώς το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας θα είναι ένα τέτοιο μέτρο Ε, αν θα μπορούσαν να, να συλλεγούν τα στοιχεία, να γίνει μια ανάκριση μέσω βίντεο διάσκεψης ή μιας προσωρινής μεταγωγής ε, με την ιδιότητα του μάρτυρα για ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα χρειάζεται να εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Υπάρχει επίση το θέμα που συζητάτε για μια ε, περιορισμού του χρόνου κράτησης πριν την ε, εκδίκαση της υπόθεσης. Μια απόφαση η οποία εκκρεμεί για, τις χρηματικές, ε, για τα χρηματικά πρόστιμα, επίσης η δυνατότητα να εκτεί την ποινή του υπόθεση με περιοριστικού όρου στο κράτος το οποίο βρίσκεται χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κράτος που υπέβαλε την ποινή ένα κρατούμενος ο οποίος ε, καταδικάστηκε ερήμην. Αυτά είναι κάποια από τα μέτρα που ευτυχώ διαπιστώνω ότι η κυβέρνηση συνεργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, τα έχει συμπεριλάβει και θα προσπαθήσει να τα να έρει το opt-out, να αρχίσει να τα εφαρμόζει. Δυστυχώς το θέμα της έκτησης ποινής υπό περιοριστικούς όρους δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Ε, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος γιατί δεν είναι λογικό ε, να εφαρμόζουμε τα άλλα χωρίς ε, το, το θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα μέτρα νομίζω θα μπορούσαν κάπως να μειώσουν την κατάχρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που γίνεται Επομένως, ε, η στρατηγική απόφαση που θα πρέπει να πάρουν οι σκιώδεις εισηγητές, και ολοκληρώνω, η στρατηγική απόφαση λοιπόν που πρέπει να πάρουμε είναι αν πρόκειται να απευθύνουμε έκκληση για νομοθετικές αλλαγές ή θα απευθύνουμε έκκληση να ανοίξει το ευρωπαϊκό έντελμα Σύλληψη εκ νέου και να τροποποιηθεί ή αν θα μιλήσουμε αν θα καλέσουμε για οριζόντια μέτρα αμοιβαία αναγνώριση ή για ανάληψη δράση, ε, για να καλυφθούν κάποια κενά όπω ε, για την προφυλάκηση και τι συνθήκε κράτηση. Υπάρχει κάποια νευρικότητα για το να ξανανοίξει το Ευρωπαϊκό Δελμα ε, και να οπισθοδρομήσουμε σε παλιές καθυστερήσεις έκδοσης. Όμως φυσικά στο εγγύης μέλλον και η συγγήτρια και οι σκιώδεις συγγητές θα πρέπει να επικεντρωθούν για το τι ακριβώς θέλουν να ζητήσουν. Ευχαριστώ κυρία Λάτφορτ για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας ε, και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους Κιώδης. Παρακαλώ, κυρία Καλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από δύο συναντήσεις των σκιωδών συγητών μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση της συγκητρίας τις ερωτήσεις και τα προβλήματα που έχουν τεθεί από την κυρία Λάτφορτ. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα προβλήματα αυτά. Και αν δούμε τα δεδομένα, τα στοιχεία για το πώς χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ποιες αποκλήσεις υπάρχουν μεταξύ των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί και όσων εκτελούνται, είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα για το σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή αυτού του Ευρωπαϊκού Ενταλματο Σύλληψη σε ορισμένα κράτη-μέλη ή μπορεί να χρησιμοποιείται δυσανάλογα σε κάποια άλλα κράτη-μέλη. Και μπορεί να πρέπει να καλυφθούν για κάποια κενά όχι μόνο στο θέμα της εφαρμογής, αλλά και στην απόφαση πλαίσιο. Στη δεύτερη συνάντησή μας ε, συζητήσαμε τα σημεία στα οποία θέλουμε να επικεντρωθούμε. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε τα θέματα αυτά με την εισηγήτρια και θα συνεχίσουμε όλο μας το έργο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε το θέμα του ελέγχου της αναλογικότητας. Γιατί θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις αποκλήσεις Μπορεί να χρειαζόμαστε να πληρείτε μία συγκεκριμένη λίστα αντικειμενικών κριτηρίων από το κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος, αλλά εξετάζοντας τα διάφορα έγγραφα και μέσω και της ακρόασης που οργανώθηκε από τους φιλελευθέρους, είδαμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να έχουμε έναν ε, διπλό έλεγχο της αναλογικότητας, δηλαδή να ελεγχθεί ένας κατάλογος κριτηρίων σε σχέση με το έντελμα και από τα δύο κράτη. Επίσης, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που μπορεί να τεθεί από εμά και θα πρέπει να συζητηθεί εδώ, είναι το θέμα της απόσυρσης ε, του εντάλματος από το κράτος έκδεσης, αν ε, το κράτος το οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνηθεί να το εκτελέσει αν δεν πληρούνται τα αντικειμενικά κριτήρια. Το τρίτο μεγάλο πακέτο είναι οι διαφορές στα οικονομικά δικαιώματα μεταξύ των κρατών μελών και πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί γιατί είδαμε ότι η προφυλάκηση είναι, διαφέρει σε ό,τι αφορά το χρόνο και φυσικά διαφέρουν και τα γεγονότα στα κράτη-μέλη. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε κάποια πολύ σημαντικούς τομείς, κάποια πολύ σημαντικά θέματα σε αυτή την έκθεση και υπογραμμίζω ότι συμφωνώ ότι συμφωνώ με αυτά τα μεγάλα προβλήματα που απαριθμήθηκαν προηγουμένως από την κυρία Λάτφορτ. Κυρία Σίπελ, επίσης και Όδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συγγήτριά μας, Σάρα Λάτφορντ, πολύ εμπεριστατωμένο μας περιέγραψε την όλη συζήτηση και νομίζω μέχρι τις ε, συναντήσεις ε, μέχρι τώρα συζητήσαμε δύο βασικά θέματα. Πρώτον, ότι βασικά η ιδέα αυτή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης ε, είναι καλή, είναι θετική, γιατί θέλουμε να ε, προσφύγουν ε, στα δικαστήρια πολύ σύντομα κατά των παραβατών σημαντικών εγκλημάτων. Και βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεταφορά αυτού του μέτρου, τα οποία δεν έχουν λυθεί όλα και πρέπει να τα εξετάσουμε ε, λεπτομερώς. Η Σάρα Λάτφορντ ανέφερε και η συνάδελφος μου ε, κυρία Γκάλ ανέφερε επίσης μερικά ειδικά ε, σημεία και θα περιοριστώ στις βασικές, στα βασικά στοιχεία που νομίζω ότι είναι τα σημαντικότερα. Καταρχάς, οι συνθήκες κράτησης. Εδώ πιστεύω ότι σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι συνθήκες είναι προβληματικές. Πρέπει να εξετάσουμε και πέραν του ευρωπαϊκού εντάλματος ε, πώς, ε, πώς είναι οι συνθήκες αυτές, ε, ιδιαίτερα στις, στην προδικαστική κράτηση και ποια είναι τα minimum standards, τα οι μίνιμουμ, οι ελάχιστες συνθήκες τις οποίες, οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της προφυλάκησης ε, η οποία μπορεί να είναι ε, πολύ μακρά, ε, πρέπει να δούμε πότε θα αρχίσει η δικαστική διαδικασία. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ύποπτα εγκληματικών πράξεων, αλλά ποινικών αδικημάτων μάλλον, που όμως κρατούνται επί μακρό χρονικό διάστημα προφυλακισμένοι χωρίς να αρχίζει η δικαστική ε, διαδικασία και ε, πολλές φορές τα άτομα αυτά ξεριζώνονται από το ε, καθημερινό τους περιβάλλον, από τη δουλειά τους, από την, απομονώνται από τις οικογένειές τους και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις και επίσης επιπτώσεις κόστους που δεν θα έπρεπε να σημειώνονται καθόλου. Είναι ε, λοιπόν σημαντική εξέταση αυτών των συνθήκων κράτησης. Έχουμε επίσης το πρόβλημα ότι έχουμε πολύ διαφορετικές ε, ε, δικαστικές νομοθεσίες στα κράτη-μέλη, δικαστικές διαδικασίες. Αρχίσαμε την επεξεργασία του κοινού οδικού χάρτη, αλλά ακόμα δεν έχουμε επιτύχει την εξομοίωση. Μόλις έχουμε υπερψηφίσει το δικαίωμα ε, του, της υπεράσπισης, επίσης ε, το, την κάλυψη του δικαστικού κόστους, του κόστους της δικαστικής διαδικασίας και ε, πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτές οι αποφάσεις που έχουμε λάβει θα βοηθήσουν στην διευθέτηση των εκκρεμών προβλημάτων του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Όσον αφορά τώρα τη σημασία του ευρωπαϊκού εντάλματος αλλά και τα προβλήματά του, βεβαίως από τη μία έχουμε τις βασικές αρχές και ε, από την άλλη πλευρά έχουμε μία ευρεία σύμπτωση απόψεων για την ε, λειτουργία, για την ε, εφαρμογή του. Και επίσης όλοι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα και ειδικά ε, στο, εκεί όπου γίνεται, αρχίζει η δικαστική διαδικασία. Το θέμα είναι ότι θα προετοιμάσουμε μία έκθεση νομοθετικού περιεχομένου που όμως θα αφήσει ανοιχτά άλλα, άλλες πτυχές τις οποίες θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε Πρέπει λοιπόν να δούμε εάν αυτά τα εκκρεμή ζητήματα θα τα καλύψουμε στην έκθεση για, την, για το ευρωπαϊκό ένταλμα ή αν θα χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα νομοθετικής φύσεως όπου μπορούν να καλυφθούν αυτές οι εκκριμότητες. Ε, μετά από τη συζήτηση που θα κάνουμε όλων αυτών των προβληματικών θεμάτων θα καταλήξουμε σε μία απόφαση. Βασικά όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία έκθεση νομοθετικού περιεχομένου και προσβλέπω με χαρά, με ικανοποίηση την ε, μελλοντική συζήτηση την οποία θα κάνουμε με, την, ε, με τον εισηγητή και τους κοιόδους εισηγητές. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ να προχωρήσουμε με τους βουλευτές που θέλουν το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Όπως ε, είπατε, η απόφαση πλαίσιο του 2002 έχει δεσπίσει ένα βασικό μηχανισμό για την εφαρμογή και την προαγωγή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης ε, οι θύνοντες ε, φυσικά ο χειρότερος εχθρός είναι η κατάχρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και η προσφορά πολιτικής προστασίας από κάποιους. Ε, και από την άλλη έχουμε δει ότι υπάρχει πολιτικοποίηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη σε ορισμένε περιπτώσεις. Συμφωνώ όμως, υπόθηκαν λοιπόν από συνάδελφο για ε, το διπλό έλεγχο της αναλογικότητας και στα δύο Αλλά θα πρέπει να καλύψουμε τα παραθυράκια που υπάρχουν, ε, το χάρη όταν ε, η Γερμανία εξέδωσε ε, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ε, για τον επικεφαλή της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ιουκοσλαβίας στην Κροατία και πριν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νομοθεσία προκειμένου να αποφευχθεί η σύλληψη του ατόμου αυτού και η έκδοσή του. Και τώρα, σε συνεργασία με την Κομισιόν, για να το πούμε διπλωματικά, μιλώντας για συνεργασία, το Κοινοβούλιο της Κουρατίας ε, τελικά άλλαξε αυτό το νόμο, αλλά και υπάρχει τώρα και νέα προσπάθεια να τροποποιηθεί το Σύνταγμα προκειμένου να αποφευθεί αυτή η έκδοση. Και υπάρχει πολιτική πίεση στην εισαγγελία για να δικαστεί ο άνθρωπος αυτός ε, στην Κροατία. Και έτσι θα συνεχιστεί μια δικαστική διαδικασία στην Κροατία για να αποφευκτεί η έκδοση στα γερμανικά δικαστήρια. Τελικά, αν τα μεταφράσουμε σε πολιτική γλώσσα όλα αυτά τα δικαστικά παιχνίδια, μιλάμε για παροχή πολιτικής προστασίας για κάποιον που κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα. Στην αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και ε, στα κράτη έκδοσης ε, αλλά και στις χώρες στις οποίες απευθύνεται το αίτημα που θέλουν να προσφέρουν πολιτική προστασία προκειμένου να ασκήσουν πολιτική πίεση στα δικοστήρια που θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μωρές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η κυρία Λάτφορτ ε, με μεγάλες λεπτομερίες έκανε την παρουσίασή της και αυτό είναι μια ένδειξη για το πώς θα προχωρήσει η αναθεώρηση. Και οι σκιώδεις έχουν προχωρήσει με ένα πολύ καλό τρόπο, γιατί η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντέλματος σύλληψη θα εξεταστεί σε όλο το Κοινοβούλιο. Το ένταλμα σύλληψης νομίζω έχει γίνει ε, συμβολικό όλης, ε, όλου του τομέα της ποινική δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων θεωρείται ως ακρογωνίας λήθος και είναι συμβολικό για το πώς λειτουργεί όλος ο τομέας αυτός ε, και όχι μόνο λόγω της Βασιλείου. Νομίζω ότι η αναθεώρηση θα είναι σημαντική για όλους και θα πρέπει να υλοποιηθεί με έναν λεπτομερή τρόπο. Νομίζω ότι η κυρία Λάτφορτ αυτό ακριβώς κάνει. Αλλά το διακύβευμα εδώ είναι ότι πρέπει το σύστημα έκδοσης να λειτουργεί. Παραδείγματος χάρη, οι αναθεωρήσεις που έχουν δημοσιευτεί μας δείχνουν ότι βασικά λειτουργεί το ένταλμα, αλλά χρειάζεται μεταρρύθμιση. Και το μέγεθος της μεταρρύθμισης αυτή θα έχει να κάνει με μια αξιολόγηση που θα γίνει από αυτό το Κοινοβούλιο για το πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψη. Ήσαν ε, ανέφερε για ε, τελικά ποιε αλλαγέ θα χρειαστούν, αν θα είναι νομοθετικέ αλλαγέ ή οριζόντιου τύπου ή αν θα καλύψουμε τα κενά. Και αυτό θα είναι η τελική δοκιμασία για το πώς ε, θα αλλάξουμε το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα πολύ προσεκτικά. Η έλλειψη της αναλογικότητας ε, και οι μακρές περίοδοι προφυλάκησης, ε, οι συνθήκες φυλάκησης, όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε και να τα δούμε πολύ προσεκτικά. Γιατί Είχαμε πάρα πολλές ιστορίες στον τύπο σε πάρα πολλές χώρες ε, και νομίζω ότι η κυρία Λάτφορ είναι το κατάλληλο άτομο που μαζί με του Κιώδη θα προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν ε, τις ιστορίες στον τύπο από την αντικειμενική πραγματικότητα. Είχαμε και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με ακαδημαϊκούς και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να προταθούν εδώ και νομίζω ότι ε, μία από τις ε, μεγάλες ελευθερήσεις ε, που είχαμε στην, στον τομέα ΔΕΗ είναι ακριβώς αυτή. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα μεγάλο διακύβευμα και χαρακτηριστικά η κυρία Λάτφορτ μας παρουσίασε μια πολύ λεπταμερή πρώτη ανταλλαγή αποψη Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργεί σωστά η αναλογικότητα και όταν τελικά έχουμε, είμαστε σίγουροι ότι είναι καλό το σύστημα του Ευρωπαϊκού της Σύλληψης και λειτουργεί, θα είμαστε, και λειτουργεί, θα είμαστε σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ κύριος Μπρόνς. Πολλές φορές οι αντιρρησίες είναι και εκείνοι που είναι εναντίον της έκδοσης. Εγώ δεν είμαι καθόλου εναντίον της έκδοσης. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα πρέπει να εκδοθούν. Όσον αφορά τώρα την την, το ευρωπαϊκό ένταλμα ως ευρωπαϊκό μέσον. Εγώ είμαι αντίθετος, αλλά είμαι και αντίθετος επί της ουσίας, διότι το ε, δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να το αρνηθεί επειδή δεν υπάρχουν ε, μάρτυρες. Πριν εισαχθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, οι δικαστές ε, στη χώρα μου θα έπρεπε να είχαν πολύ σοβαρές ενδείξεις και εν συνεχεία αποδείξεις για την ενοχή του κατηγορούμενου. Ε, Βεβαίω η διαδικασία ώσπου να συλλεχθούν όλα αυτά τα στοιχεία ήταν χρονοβόρα, αλλά πολλές φορές η δικαιοσύνη αργεί. Τώρα, όσον αφορά τη χώρα η οποία ζητάει την έκδοση ενός ατόμου, εκεί το αδίκημα του θεωρείται ε, ποινικό, ενώ στη χώρα όπου διαμένει κατοικεί, δεν, ε, στη χώρα διαμονής του δεν θεωρείται αδίκημα η πράξη του. Ε, γι' αυτό και εγώ είμαι αντίθετος στο ευρωπαϊκό ένταλμα και όσο υπάρχει αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ισχύει και για το Ενωμένο Βασίλειο, ε, για να είμαι δίκαιος, θα προτιμούσα το ευρωπαϊκό ένταλμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος να προηγείται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας, έτσι ώστε να αποφύγουμε δαπανηρές και χρονοβόρες ε, προσφυγές. Ευχαριστώ. Κυρία Ρόμερο Λόπες, ευχαριστώ. Ναι, πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη είχε εντοπίσει στην έκθεση της τις αναλογίες που υπάρχουν για το έντελμα σύλληψης και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λάτφορτ αν ε, πράγματι έγινε μια μελέτη αυτής της ε, τυπολογίας ε, για τα πλημελήματα τα οποία ε, εκδόθηκαν ε, εντάλματα σύλληψης ευρωπαϊκά και προκλήθηκε αυτή η έλλειψη αναλογικότητας γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ε, είχαμε πολύ αρνητικό αποτέλεσμα όταν είχαμε δυσανάλογη χρήση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αυτή, λοιπόν, αυτός ο ορισμός των πλημελημάτων θα έπρεπε να πλαισιωθεί περισσότερο, να γίνει πιο συγκεκριμένος ορισμός. Και πράγματι αυτό που συμβαίνει με τη μεταρρύθμιση είναι ότι την κάνουμε ενδιάμεσα, όταν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο δικός χάρτης σε σχέση με τις δικονομικές εγγύσεις. Και είναι προφανές ότι δεν έχουμε συζητήσει το θέμα των συνθήκων κράτησης, ούτε την δωρεάν νομική συνδρομή. Και Όντω, υπάρχουν κάποιες βελτιώσει, περνώντα χάρη σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, δηλαδή να υπάρχει πρόσβαση σε δικηγόρο, στην υπεράσπιση τόσο στο κράτος έκδοσης όσο ε, και στο κράτος εκτέλεσης. Όμως παραμένουν κάποια σημαντικά θέματα όπως οι συνδικές κράτησης, ο χρόνος κράτησης και η δωρεάν νομική συνδρομή. Γιατί όπως είπε και η συνάδελφος Σίπελ μπορεί να προκύψει εξή περίπτωση, να γίνει ένα λάθος, να μην υπάρχει δυνατότητα προσφυγής, να μην αναλάβει κανείς την ευθύνη, να πρόκειται για πλημέλημα, να έχει περάσει ο ύποπτος πάρα πολύ χρόνο στη φυλακή και νομίζω ότι όλα αυτά θα έπρεπε να τα αποφύγουμε. Αυτή η αναθεώρηση θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Και υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα που θέλω να τονίσω, γιατί δεν ξέρω αν οι συγγητρικές και οι συγγητές ε, έχουν συζητήσει αυτό το θέμα. Όταν ε, ο ορισμός του σοβαρού εγκλήματος που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης χρησιμοποιείται ως βάση για άλλες οδηγίες που έχουμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο, παραδείγματο χάρη για το PNR των επιβατών υπάρχουν ε, ορισμένα ε, αδικήματα που θα έπρεπε να αναθεωρηθούν όπως παραδείγματο χάρη η βοήθεια στους λαθρομετανάστες. Και είδαμε τι συνέβη στη Λαπεντούσα, επομένως πρέπει να αναθεωρήσουμε πραγματικά αυτό τον καταλόγο των 132 δικημάτων γιατί αν το λάβουμε αυτό ως βάση, αυτό το αδίκημα τώρα έχει τελώς διαφορετική αντίληψη σε σχέση με την στιγμή κατάρτισης εκείνου του καταλόγου των 132 δικημάτων γιατί έχουμε τώρα το αδίκημα της εμπορίας ατόμων, της εμπορίας ανθρώπων. Επίσης έχουμε το αδίκημα που ε, είναι προφανές ότι θα έπρεπε να καταργηθεί, γιατί δεν έχει νόημα σε ένα κατάλογο σοβαρών εγκλημάτων που κατόπιν χρησιμοποιείται ως βάση για άλλες οδηγίες. Και θα εκμεταλλευτούμε για να καταθέσουμε τροπολογίες και για άλλα θέματα που έχουν ήδη τονιστεί και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ. Κύριος Κίκοφ θέλει να παρέμβει πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν και μετά ε, στον εισηγητή. Ο κύριος Κίκοφ, λυπάμαι που ε, έπρεπε να φύγω από την αίθουσα για λίγο, αλλά ήθελα να κάνω μερικές ε, σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, θέλω να είμαστε σαφείς ότι το μέσον αυτό, το ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι πολύτιμο για σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης. Ε, επίσης, είναι ένα σημαντικό μέσον διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα ταχύτατα, ιδιαίτερα μετά την ε, ε, διάσταση των συνόρων του, του Σέγγεν και των κενών που σημειώνονται, αλλά ε, πρέπει να πω επίσης ότι πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι εδώ βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και πρέπει να αναθεωρήσουμε το όλο πλαίσιο επειδή υπάρχουν προβλήματα όπως η αναλογικότητα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα αναλογικότητας και να εισαχθεί στο μέσον αυτό για να αποφύγουμε ορισμένα λάθη του παρελθόντος πρέπει να ορίσουμε ε, έναν κατάλογο αδικημάτων ε, και την, ε, σύμφωνα με τις ερμηνείες στα κράτη-μέλη και τον τόπο του αδικήματος όπως σημειώνεται το αδίκημα. Επίσης, πιστεύω ότι είναι σημαντικά να, δοθούν εγγυήσεις και να υπάρχουν περιορισμοί ε, όπως και να τονίσουμε περισσότερο τα πλεονεκτήματα του ευρωπαϊκού εντάλματος. Ε, ε, ε, έχουμε δει ορισμένα ωφέλη, όμως τώρα χρειάζεται μία, μία μεταρρύθμιση για το ευρωπαϊκό ένταλμα, αλλά γενικά βασικά το ένταλμα αυτό αποδείχθηκε πολύ ωφέλιμο και ευχαριστώ την εισηγήτρια που δέχτηκε να προχωρήσει το όλο θέμα. Thank you very much, Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο που αυξάνει και ωφελεί την δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και επιδιώκει να συμβάλλει στην επίστευξη του, του ενός πολύ βασικού στόχου της ποινική δικαιοσύνης, την αποφυγή της, ε, Επίσης πιστεύω ότι το μέσον αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της δικαιοσύνης και ενισχύει και την εμπιστοσύνη μεταξύ μας στα δικαστικά συστήματα. Ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια που διοργάνωσε μία η μερίδα πριν από δύο εβδομάδες ε, με το θέμα του ευρωπαϊκού εντάλματος και όλα αυτά που συζητήθηκαν ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να προβάλλουμε την θέση της ε, Κομισιόν όσον αφορά τις νομικές δυνατότητες ε, το 2014 και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης σε κρατικό επίπεδο. Γι' αυτό θα ήθελα και μέσα στο πλαίσιο των διαδικασιών κυρώσεων μέσα στο πλαίσιο της μεταφοράς σε εθνικά δίκαια, θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν αν έχει αλλάξει ε, τους λόγους ε, για την ε, μη εφαρμογή της, του εντάλματος. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν έχει αλλάξει την τοποθέτησή της η Κομισιόν όσον αφορά την επιβολή νομικών μέτρων σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν θέλει να εφαρμόσει τις ε, διατάξεις ε, του εντάλματος. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν πώς θεωρεί το ένταλμα αυτό μέσα στο πλαίσιο της γενικής δικαιοδοσίας των κρατών μελών. Υπάρχει περιθώριο κατάχρησης ε, της χρήσης, κατάχρησης του εντάλματος αυτού μέσα σε ορισμένα δικαστικά και δικονομικά πλαίσια. Και όταν είχε αποφασιστεί το ένταλμα τότε, ε, είχαμε θέσει μία επιφύλαξη και είχαμε πει ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα δεν θα εφαρμοστεί για ποινικά δικήματα τα οποία έχουν γίνει πριν από το 2004. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά νομικά θέματα τα οποία πιστεύω εάν απαντηθούν θα συμβάλλουν σε μια καλύτερη και σαφέστερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος. Εγώ γενικά υποστηρίζω θερμά το ευρωπαϊκό ένταλμα και έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για την λειτουργία της διαδικασίας έκθεσης και της ε, συνεργασίας της δικαιοσύνης μεταξύ των κρατών μελών της ποινικής δικαιοσύνης. Μάλιστα. Θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και στην Κομισιόν ε, και να πάρει το λόγο και η συγγήτρια. Οπότε με μακρηγορήσετε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια για τη λεπτομερή παρουσίασή της. Και όπως είπε και ο κύριος Μωράες, το σύστημα έκδεσης πρέπει να λειτουργήσει, αλλά συμφωνώ με ορισμένου από τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να γίνει αυτό χωρίς να πολιτικοποιείται αυτό το σημαντικό εργαλείο ε, που έχει ανοίξει και ένα, μια πόρτα στα θύματα που είναι θύματα όχι μόνο εγκλημάτων και οργανωμένων εγκλημάτων αλλά και πλημελημάτων που μπορεί να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ζητώ από την εισηγητρία και τους κοιόδης να λάβουν υπόψη και τα δικαιώματα των ε, θυμάτων, ε, να μην παραβιάζονται λόγω της διαφορετικότητας στις διάφορες εθνικές νομοθεσίες. Ε, και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Τέλμα Σύλληψης είναι ένα μέσο που πρέπει να βελτιωθεί, αλλά πάντοτε να χρησιμοποιείται για την κατάλληλο σκοπό. Και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνεται σε ό,τι φορά το θέμα της αναλογικότητας του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο η κυρία Τρίσα Χάρκιν. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα εκ μέρους της Κομισιόν να πω ότι καλωσορίζουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Η Κομισιόν ε, παρακολούθησε και την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση που την προείδρευσε η κυρία Λάτφορτ και οργανώθηκε από το Άλντε πριν δύο εβδομάδες περίπου. Η συζήτηση αυτή αντικατοπτρίζει και τα σχόλια σήμερα το πρωί και ήταν μάλλον και σε πιο τεχνικό επίπεδο. Εμεί παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον ε, το έργο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και γνωρίζουμε την παράλληλη μελέτη που υλοποιεί η Κομισιόν και έχουμε προγραμματίσει να συναντηθούμε και με τους ακαδημαϊκούς ε, αλλά και τους νομικούς για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν ε, αναφερθεί εδώ και η Κομισιόν τα γνωρίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες. Αλλά να σας πω ότι εκ μέρους της Κομισιόν ενθαρρυνόμαστε από την επικοδομητική και ρεαλιστική προσέγγιση που ακολουθεί η και σκιώδης συζητητής ε, στο να προσεγγίσουν τα δύσκολα ζητήματα και τα σημεία όπου βλέπουμε μία ευρύτερη εικόνα ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληξης δεν υπάρχει στο κενό έχουμε μία σειρά μέτρων και τα μέτρα των οικονομικών δικαιωμάτων που το, που το συμπληρώνουν, αλλά και τα υπόλοιπα μέτρα αμοιβαία αναγνώριση. Ε, και θέλω να αφαιρθώ σε ερωτήσει του κ. Πρόκοβιτ. Νομίζω ότι συζητήθηκαν και στην ακρόαση των ε, φιλελευθέρων, όμως το θέμα της ε, εφαρμογής πρέπει να συζητηθεί. Έχουμε και πολλά άλλα συμπληρωματικά μέσα που δεν έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη και αν ήταν διαθέσιμα τώρα στους πολίτες θα έδιναν πάρα πολλές εναλλακτικέ για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Τώρα δεν θα πάω παραπέρα. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλη αυτή τη δουλειά. Θα συνεισφέρουμε που είναι δυνατό και θα συναντηθούμε με τους ε, αρμόδιους που υλοποιούν τη μελέτη και φυσικά εκτιμούμε την επικοδομητική και λεπτομερή δουλειά της εισηγήτριας και των σκιωδών. Και σε πάλι εσείς κύριε Λάτφορτ για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους ε, που παρανέβησαν, όλους τους σκιώδεις τους ε, ευχαριστώ προσωπικά και για την υποστήριξη που εξέφρασαν και τις προτάσεις τους. Νομίζω, όπως είπε και η κυρία Χάρκινς από την Κομισιόν, προσπαθούμε εδώ να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Και όπως είπα, να είμαστε αντικειμενικοί. Αν θέλετε, εγώ έχω μια εμπειρία την οποία προσπαθώ να, να, να αξιοποιήσω, η οποία είναι διαφορετική από αυτό που λέει ο κύριος Μπρόγκς. Ε, το άκουσα προσεκτικά, αλλά διαφωνώ. Εγώ καταρχήν δεν έχω καμία αντίρρηση να ληφθούν ε, μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξορισμού θαυμάσιο ή δεν μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι να βελτιώσω το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Να. Ε, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση όμως να ξαναγυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση όπου μπορούσαν οι υποπτοί να καταφεύγουν σε ορισμένα κράτη ή σε ορισμένες περιοχές και να βρισκόνται περάνω του νόμου, να παραμένουν ατιμόρυτοι εκεί. Και αυτό δεν αναφέρεται μόνο, δεν, δεν έχει σχέση μόνο με την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα, έχει σχέση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Και αυτή απειλείται όταν δεν ε, ε, προσάγονται στη δικαιοσύνη οι εγκληματίες. Προσπαθούμε όμως να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα του κατηγορουμένου και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Αυτή είναι η προσπάθεια σε οποιαδήποτε ποινικό σύστημα. Είναι λοιπόν ένα παζλ εδώ. Είναι δύσκολο το ε, θέμα και είναι μεγάλη πρόκληση να καταφέρουμε να ε, το αντιμετωπίσουμε σωστά. τελικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και του Δικαστηρίου θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα μεταγράψουν αυτή την νομοθεσία και πώς θα αξιοποιήσουν στο εθνικό τους, στην εθνική τους ένομη τάξη αυτά τα μέρα, μέτρα. Το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ακολουθήσει μια μάλλον συντηρητική προσέγγιση. Επομένως δεν έχουμε και πολλή νομολογία από το δικαστήριο για να βασιστούμε σε αυτήν. Ωστόσο, ε, είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου η αδράνεια ε, στην προσπάθεια από την πλευρά του Δικαστηρίου και της Επιτροπής να υπάρξουν κυρώσει έτσι ώστε τελικά να εφαρμοστούν τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, είτε αν αυτά αφορούν την ποινική συνεργασία, είτε αν αφορούν την ε, νέα αγορά. Είναι εξίσου απαράδεκτο να δρανούμε και στα δύο ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσπαθώ να έχω μια αντικειμενική προσέγγιση. Δεν λέω ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη είναι ε, εξορισμού τέλειο επειδή είναι ευρωπαϊκό, ούτε ότι είναι εξορισμού κατακριτέο επειδή είναι ευρωπαϊκό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να το βελτιώσουμε. Και διάφορα χρήσιμα στοιχεία άντλησα από τις προτάσεις των συναδέλφων και θα προσπαθήσω να τα ενσωματώσω στην πρότασή μου. Τελικά τι προσπαθούμε εδώ, να, να δημιουργήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ποινική συνεργασία, ποινικό σύστημα ε, απόδοσης δικαιοσύνης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα κοινό ποινικό κώδικα. Πρέπει απλώ να υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας στο δικονομικό επίπεδο, μια ε, ε, συγκρισιμότητα μεταξύ των ποινικών συστημάτων και ποινικών κωδικών χωρίς να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια πλήρους εναρμόνισης. Αυτή, λοιπόν, αυτό το εγχείρημα έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορα συγκεκριμένα στη σημεία και προσπαθούμε με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψης να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από αυτές τις εντάσεις. Θα ήθελα επίσης να πω, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και ιδιαίτερα την κυρία Κλόντια Γκοτιέρη, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με βοήθησε πάρα πολύ και όταν είχα ετοιμάσει την έκθεση για το δικαίωμα στη διαρμηνία κατά τη διάρκεια των διαδικαστικών ποινικών διαδικασιών και οι γνώσεις της ήταν πολύτιμες. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να υποφελούμαστε από αυτές τις γνώσεις. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Λάτσφορτ. Σας ευχαριστώ επίσης που ευχαριστείτε την ε, γραμματεία. και ιδιαίτερα την Κλάουδια Βαλτιέρη, η οποία πάντα μας βοηθάει εξαιρετικά πάρα πολύ οποτεδήποτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα ποινική συνεργασία, δικαστική συνεργασία. Ωραία. Κάναμε νομίζω μια διεξοδική συζήτηση που ήταν χρήσιμη και επικοδομητική όσον αφορά το κατά πόσο χρειάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Έχει έρθει η ώρα να το επανεξετάσουμε, μιας και υιοθετήθηκε το 2002 και τώρα πλέον έχει υλοποιηθεί πλέον, ε, και μπορούμε να κρίνουμε τι λειτουργήσε και τι δεν λειτουργήσε. Μπορούμε επίσης να κρίνουμε τον τρόπο που τα κράτη-μέλη μετέγραψαν την ε, απόφαση πλαίσιο και να βρούμε τρόπους να την ενισχύσουμε, όχι να την αποδυναμώσουμε. Γιατί Όπω είπαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ήταν ένα μεγάλο βήμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κικαιώνα γραφειοκρατία που είχε δημιουργήσει το παραδοσιακό σύστημα έκδοση κρατουμένων. Με τόσα πολλά προβλήματα, όχι μόνο πρακτικά, αλλά και μια φιλοσοφική σκοπιά θα έλεγα, όσον αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, ε, έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών συστημάτων και των δικαστικών αρχών, το γεγονό ότι δεν υπήρχε αμοιβαία αναγνώριση. Ε, Αντιθέτω με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, εκφράζουμε την ε, πεποίθησή μας και τη βούλησή μας να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτές τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις. Να σας ενημερώσω ότι στις 27 Νοεμβρίου θα γίνει η συζήτηση. Και επίσης ενημερώνω ότι έχουμε δημόσια ακρόαση 3 και μισή στην ίδια αίθουσα. Στις 3 θα γίνει μια ανοιχτή σύνοδος ε, του, του Προεδρίου, στην οποία καλώ τα μέλη. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν λοιπόν ε, σε αυτή, τη συνεδρία, σε αυτή την, την ανοιχτή συνεδρίαση του προεδρίου, επισημαίνω ότι θα ξεκινήσουμε μισή ακριβώς. Θα είμαι αυστηρός όσον αφορά την τήρηση του χρόνου Νομίζω το καταφέραμε καλά με την τήρηση της ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί. Η δημόσια γρόση θα ξεκινήσει στι 3.30 ακριβώ. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε αργότερα.